Πέρας της ψηφοφορίας. 13 υπέρ 13 κατά, επομένως απερίφθη η 258. 259 γκρέσλε στάς, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω πως το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, αλλά καλύτερα να επαληθεύσουμε. 259 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 12 υπέρ 14 κατά απερίφθη. 2.60 ηλεκτρονική ψηφοφορία για, το, για την τροπολογία 2.60. Πέρα τη ψηφοφορία. Απερίφθη 12 ψήφοι υπέρ, 13 ε, κατά. 2,61 και εδώ ηλεκτρονική ψηφοφορία. 2.61 ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας. Ισοψηφία, επομένως απερίφθη η τροπολογία 2.61. 2.62 ε, να κάνουμε αμέσως ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ κοντινό. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία επί της 2.62 πέρας. 12 ψήφοι υπέρ, 14 κατά, απερίφθη, λοιπόν. Η 263 έχει αποσυρθεί, 264 γκρέσλε στάς. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία επίσης. Πέρας. Ισοψηφία 13 ψήφοι υπέρ 13 κατά επομένως απερίφθη, 265 ηλεκτρονική ψηφοφορία για μια ακόμα φορά. 13, 14 verworpen en dan... Απερίφθη 13 υπέρ 14 κατά 266 ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 23 ψήφοι υπέρ 4 κατά, επομένως εγκρίνεται. 267 έχει αποσυρθεί, 268 γκρέσλι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 269 Bradford Τσαρνέσκι υπέρ κατά αποχές. Νομίζω πως έχει απορριφθεί η τροπολογία 269 να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Λοιπόν, για να δούμε. Ε, τροπολογία 269 πέρα της ψηφοφορίας. Έχει απορριφθεί 13 ψήφοι υπέρ, 14 κατά. Απερίφθη. 2,70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως συγκρίνεται. 2,70 ε, υπέρ κατά 2,71 μάλλον 2, υπέρ κατά αποχές επαλήθευση 2,79 πίπερ ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 16 ψήφοι υπέρ, 11 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 272 πίπερ πάντα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 273 Παναγιώτοβα υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 274 Ερνχάουζερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 275 Πίπερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 276 Στάση υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 277 Οντί υπέρ. Κατά. Αποχές ε, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Πολύ κοντινό να ε, κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας της, επί της 277, 11 υπέρ, 14 ψηφικά κατά, επομένως απερίφθη 278 Bradburn υπέρ κατά, αποχές, νομίζω πως εγκρίθηκε. Όχι, δεν έχετε σχόλια επί του αποτελέσματος. Προχωράμε λοιπόν. 279 οντί κατά αποχές εγκρίνεται. 280 γκάγερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 281 Μπρατμπορν υπέρ κατά αποχές Επίσης είναι πολύ κοντινό το αποτέλεσμα, καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Επί της 281, πέρα της ψηφοφορίας, 14 ψήφοι υπέρ, 13 κατά, επομένως εγκρίνεται. 282 γκρέσλε υπέρ, κατά. Αποχές, επίσης πολύ κοντινό το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. 14 ψήφοι υπέρ, 13 κατά, επομένως ενεκρίθη. 283 πίπερ, υπέρ, κατά, αποχέσα το αποτέλεσμα για μένα είναι πάρα πολύ κοντινό. Ε, λοιπόν, για να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση πέρα της ψηφοφορίας. 14 ψήφοι υπέρ, 13 κατά, επομένως εγκρίνεται. 2.84 Παναγιώτοβα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.85 Πίπερ υπέρ, κατά, αποχές. Τι να σας πω, ηλεκτρονική επαλήθευση. Γιατί φαίνεται ότι εδώ οι αγωνιστές έχουν αρχίσει και κουράζονται. Δεν σηκώνουν τα χέρια τους καλά, πέρα της πληροφορίας. 19 ψήφι υπέρ, 7 κατά, 2,86 υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία βεβαίως. Άρχεται η ψηφοφορία. 25 ε, υπέρ, μία ψήφος κατά, συγχαρητήρια στον εισηγητή, καμία αποχή και μία ψήφος κατά, όπως σας είπα προηγουμένως, συγχαρητήρια. Για να βάλουμε λίγο τάξη στη σκέψη μας και στα πράγματά μας. Τώρα θα κάνουμε ψηφοφορίες ε, στις ειδικές εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Δεν θέλει. Κυρία Γκρέσλε, ήθελα μόνο να σας πω να σας εξηγήσω την πληθώρα των τροπολογιών, γιατί εμείς ψηφίσαμε κάποιες συστάσεις στην Επιτροπή μας και λείπουν ε, αυτές από τα όσα μας προτείνει ο εισηγητής. Δεν το θεώρησα σωστό και έχω επαναφέρει εγώ τα, τις συστάσεις των εκάστοτε εισηγητών. Γι' αυτό έχουμε τόσο πολλές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Rapporteur, και κύριοι, eh, Κύριε υπάρχουν τροπολογίες τις οποίες μπορούμε να ψηφίσουμε on block. Εγώ δεν διαφωνώ. Οι άλλες πολιτικές ομάδες ε, ε, τι λένε. Ο πρόεδρος. Από την 1 έως 18 μπορούμε να τις ψηφίσουμε on block όλες αυτές τις συστάσεις. Συμφωνείτε. Επομένως θα ψηφίσουμε από κοινού 1 μέχρι 18. 1 μέχρι 18, όχι, 1 μέχρι 25, unblock. Όχι, ναι, Γιάννη, τι λες. Ε, εντάξει, 1 μέχρι 12. Καλά. Τροπολογίες 1 έως 12, λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 13. Κρέσλε, υπέρ. Κατά αποχές ε, είναι πολύ κοντινό το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 13 Γκρέσλε. Πέρας της ψηφοφορίας. 14 ψήφοι υπέρ, 10 κατά, επομένως εγκρίνεται η τροπολογία 13. Υπάρχουν άλλες που μπορούμε να ψηφίσουμε αν μπλοκ κατά την άποψή σας. Μία-μία, τι θα κάνουμε. Από τη 14 μέχρι την 25 μπορούμε, από κοινού όχι. Οι φιλελεύθεροι δεν το επιθυμούν. 14 γκρέσλε υπέρ. Κατά. Αποχές Επίσης είναι πολύ κοντινό το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 14. Πέρας της ψηφοφορία. εγκρίνεται 15 ψήφοι υπέρ 10 κατά. Προχωρούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ασκήσετε λίγο περισσότερο, να σηκώνετε το χέρι σας. Γκρέσλε 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 16 γκρέσλε πάντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως απερίφθη, αλλά καλύτερα να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 16. 16 λοιπόν. Πέρας της ψηφοφορίας. 15 ψήφοι υπέρ, 9 κατά, επομένως απερίφθη. Επομένω εγκρίνεται, συγγνώμη. Ε, τροπολογία 17 Γκρέσλε υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως εγκρίνεται. Συμφωνείτε. Ωραία. Πάμε στη 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 έχει αποσυρθεί. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ της κυρίας Γκρέσλε κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 Γκρέσλε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 Μαρινέσκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 Γκρέσλε υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. to check myself. Πέρας της ψηφοφορίας, 15 ψήφοι υπέρ, 10 κατά, επομένως εγκρίνεται. Τροπολογία 30 γκρέσλε, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 31, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 33, κανένα πρόβλημα, πολύ ωραία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν για την τροπολογία 33 πέρας της ψηφοφορίας. 13 ψήφοι υπέρ, 12 κατά, επομένως ενεκρίθη. Είχε δίκιο ο πρόεδρος. 34 υπέρ, κατά. Αποχές. Τι να σας πω, το ΕΛΚΕ έχει κουραστεί. Λοιπόν, <laughs> άρα θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση ε, και παρακαλώ εφ' να σηκώνουν πιο δυναμικά το χέρι τα μέλη του ΕΛΚ πέρας της ψηφοφορίας. 13 ψήφοι υπέρ, 12 κατά. Επομένως περνάμε στην 35 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 36 γκρέσλε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 37 γκρέσλε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 38 γκρέσλε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 γκρέσλε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 γκρέσλε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 γκρέσλε υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 42 γκρέσλι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 γκρέσλι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 γκρέσλε υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 γκρέσλε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 46 γκρέσλε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 47 ε, του υποφαινομένου υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη, 48 σταυρακάκης υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω ότι θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία Σταυρακάκη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 15 ψήφοι υπέρ, 10 ψήφοι κατά, επομένως ενεκρίθη. 49 Παπαδοπούλου υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 50 της Ιδίας υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 51 Παπαδοπούλου υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη, 52 Παπαδοπούλου υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη, 53 Παπαδοπούλου υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω πως έχει εγκριθεί, αλλά καλύτερα να επαληθεύσουμε. Τροπολογία 53 Παπαδοπούλου, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 25 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά, επομένως ε, ενεκρίθη. Βλέπω ότι πρέπει να, να ξυπνήσετε λίγο. Επόμενη τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 55 Παπαδοπούλου υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 58 υπέρ συγγνώμη, 56 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Πού είμαστε, ρωτάει ο Πρόεδρος. Στην 57 ε, Παπαδοπούλου, υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 58 Γκρέσλε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 Γκρέσλε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 γκρέσλε έχει αποσυρθεί, 61 οντί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία από 62 μέχρι 68 μπορούμε να τις εξετάσουμε από κοινού. Ναι, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία οντί 69 να δούμε. Α, θέλετε επαλήθευση από τις τροπολογίες 62 μέχρι 68. Πολύ ωραία. Ηλεκτρονική λοιπόν ψηφοφορία. Εντάξει, πέρας της ψηφοφορίας. Να δούμε το αποτέλεσμα. 14 ψήφοι υπέρ, 12 ψήφοι κατά, επομένως ενεκρίθησαν αυτές οι τροπολογίες. Τροπολογία 69 μέχρι 71, οντί από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική. Πέρας της ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα, 18 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά, 6 αποχές. Συγχαρητήρια. And now, what do we have now? We hebben dat goed gedaan. We, hebben 12, we zijn 12 minuten voor. Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ καλά. 12 λεπτά νωρίτερα από ό,τι είχαμε υπολογίσει. Δεν είναι Μιλάνο Σαρέμο, έτσι, σαν την ποδηλατική ε, κούρσα. Ερχόμαστε στο 5 για το ευρωπαϊκό, τα ευρωπαϊκά μάλλον ταμεία ανάπτυξη στον πληθυντικό. Είναι έκθεση του κυρίου Σόντεργαρτ. Θέλει να πει τίποτα ο εισηγητής. Όχι. Ωραία. Πάμε, έχουμε τον κατάλογο ψηφοφορίες μας. ik ga mijn eigen lijst nemen. Και εγώ το δικό μου. EDF, πάμε. Ik stel voor dat we, we, we hebben de agenda aangenomen, mevrouw Ja, εγκρίναμε την ημερήσια διάταξη, δεν κάνατε κανένα σχόλιο, δεν ζητήσετε να αλλάξει. Ε, ακολουθούμε τη σειρά λοιπόν που έχουμε ορίσει στην ημερήσια διάταξη. Εντάξει, ε, ε, πρόταση λοιπόν για απόφαση ε, για απαλλαγή, ναι ή όχι. Παράγραφος 1, τροπολογία 2 Σόντεργαρτ, που προτείνει να δοθεί η απαλλαγή. Ψήφι υπέρ της τροπολογίας 2 του κυρίου Σόντεργαρτ κατά εγκρίνεται. Άρα οι τρία Έπινγκ ε, και Μπράντμον καταπίπτει και ερχόμαστε στην τροπολογία 1 Μακοβέη και Γκρέσλε είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική λοιπόν τώρα ψηφοφορία για την πρόταση. Πέρας. Εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ, 2 κατά. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε στο κλείσιμο των λογαριασμού. την 5 και την 6 δεν τις ψηφίζουμε, διότι δώσαμε απαλλαγή και πάμε στην 4, μέσως Μακοβέη Γκρέσλε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Και εδώ ηλεκτρονικά θα πρέπει να ψηφίσουμε ε, αυτό το τμήμα της απόφασης. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία έχει αρχίσει. Πέρας. 24 υπέρ 2 κατά επίσης εγκρίνεται. Τώρα έχουμε ε, το ψήφισμα. DV1 ψήφι υπέρ της πρώτης απολογίας της Επιτροπής Ανάπτυξης. Κατά αποχές εγκρίνεται. Όλε Σμιτ 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 Γκρέσλε υπέρ. Ορίστε. 20 Γκρέσλε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 3 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 γκρέσλε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύε 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύε 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 σε δύο τμήματα, τη Σουζάνα Μπζομποχάτα είμαι πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά στο ελέγξουμε παρακαλώ. Το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 22. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε. 7 υπέρ 19 κατά απορρίπτεται. Αυτό τι σημαίνει, ότι καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. Όχι. Το ψηφίζουμε. Στην 22 λοιπόν ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 όλες μίτ. υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 δρέσλε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 της κυρίας Προσμποχάτα υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται 26 της ιδίας υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 24. Το ΕΛΚ έχει ζητήσει κατά ψηφοφορία. Για την παράγραφο 24 την ψηφίζουμε ξεχωριστά. Υπέρ λοιπόν. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά χρειάζεται έλεγχο. Ψηφίζουμε λοιπόν χωριστά την παράγραφο 24. Πέρα τη ηλεκτρονική ψηφοφορία. 17 υπέρ 10 κατά. Ε, εγκρίνεται. Παράγραφος 25, τροπολογία 28, όλε μιτ σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 27 Γκρέσλε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 Όλε Σμιτ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το 30 Όλε Σμιτ. Όπως τροποποιήθηκε προφορικά. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 Όλε Σμιτ έχει ζητήσει ψηφοφορία κατά τμήματα, είπε, του πρώτου, κατά, αποχές, στο δεύτερο τμήμα, το πρώτο εγκρίθηκε, είπε κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32. Όπως τροποποιήθηκε προφορικά από τον εισηγητή, είπε κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, η τροπολογία παριθμών 33 της κυρίας Μπροσβοχάτα υπέρ. Κατά άποχες. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Δεν διαμαρτύρεστε, ωραία. Τι θέλετε, ελεγχώ. Ωραία, ελέγχουμε την 33 ηλεκτρονικά λοιπόν. Πέρας. 12 υπέρ, 15 κατά, απεριφθεί όντως. Πού ήμασταν τώρα, στην 33. Πάμε στην 34, τι ιδίε. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35, όλοι Σμίτ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37, όλοι Σμίτ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και εδώ τελειώνουν οι τροπολογίες του Όλου Σμιτ όπως και το Όλου Σμιτ Show 39 επέ κατά αποχές εγκρίνεται 40 Όλου Σμιτ κατά αποχές εγκρίνεται ΔΕΒ 2 κατά αποχές εγκρίνεται 41 όλοι Σμιτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 όλοι Σμιτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 Μακοβέι Γκρέσλε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 Τόιρα 44 Μιχαήλ Τόιρος 44 όπως φορικά τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 όλοι Σμιτ υπέρ. Υπέρ είπα. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 Μαρκοβέη Γκρέσλε. Ορίστε. Έλεγχο θέλετε για τις 45 του Όλε Σμιτ. Έλεγχος ηλεκτρονικός. 19 υπέρ, 8 κατά εγκρίθηκε. Η 46 Μάκοβέη Γκρέσλε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 Μακοβέη Γκρέσλε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεβέ 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 Λεσμίτ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία τώρα. Όχι, θέλετε έλεγχο για τις 48, ωραία. Ηλεκτρονική επαλήθευση κατόπιν αιτήματος της κυρίας Γκρέσλε. Πέρας, 10 υπέρ, 16 κατά, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία D. Του κυρίου Σόντεργαρτ, πρέπει να την ψηφίσουμε αυτή. Στην παράγραφο 5. Ναι. Ωραία. Ψηφίζουμε την τροπολογία αυτή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 μακουβέι Γκρέσλε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 Γκρέσλε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 γκρέσλε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 Σόρντεγκαρτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 Σμιτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ. Καλά. Ελέγχουμε τη 53 ηλεκτρονικά. Πέρασε. 4 υπέρ, 23 κατά. Δηλαδή πόσο λάθος μπορεί να κάνει κανείς. Ε, 54. Κανονικά στην Ολομέλη εδώ ξεσπάνε στα γέλια, αλλά είμαστε σε πιο στενό κύκλο. Ε, 54 υπέρ. Συγγνώμη. Ποιο θέλει το λόγο. Σταματάμε την ψηφοφορία. Ναι, οκ. Ε, Όχι, λάθο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 54, όλες μη υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 55, όλε μη υπέρ. Κατά. απόχέ. 56 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 Μακοβέη Γκρέσλε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 Όλε Σμιτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 7 της Επιτροπής Ανάπτυξης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 Όλε Σμιτ υπέρ κατά, Αποχέ εγκρίνεται. 8 Μακοβέη Γκρέσλε υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. 9 Όλε Σμιτ υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. 10 Όλε Σμιτ υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. 11 Όλε Σμιτ υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. Δώδεκα όλε. μη, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13 όλες μη τυπέ, κατά αποχές απορρίπτεται. 14 όλες μη τυπέ, κατά αποχές εγκρίνεται. 15 όλες μη τυπέ, κατά αποχές εγκρίνεται. 16 μακόβέ γκρέσλι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 17 μακοβέ γκρέσλι κατά αποχές εγκρίνεται. 18 μακόβέ γκρέσλι κατά αποχές εγκρίνεται ερχόμαστε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Πέρα τη ηλεκτρονική ψηφοφορία 24 υπέρ 3 κατά χωρί αποχέ. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά και σε όλου του υπολείπου που συνεισέφεραν σε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην απαλλαγή του Κοινοβουλίου Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάτι ήθελα να διευκρινίσω. Στον κατάλογο ψηφοφορία έχει παρισφρήσει ένα λάθο στο σημείο 44 στην προφορική τροπολογία τη κυρία Γκρέσλε. Φαίνεται αρνητικό πρόσημο ενώ εγώ είμαι υπέρ. Είναι τυπογραφικό μάλλον. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω στο σημείο 44, αντί για πλήν να βάλουμε ένα συν. Ευχαριστώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Της εισηγητρίας. Και ταυτόσημη του κύριου Ιβαν, υπέρ. Ένα και τρία. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Άρα, οι δύο, η τροπολογία 2, Έπινγκ, Τσαρνέκη, Τσέσκοβα, Μπράντμπορν, εκπίπτει ηλεκτρονική ψηφοφορία το πρώτο μέρος, αυτό το μέρος της απαλλαγής ε, του Κοινοβουλίου. Κλείνω την ψηφοφορία. Ψήφι 25 υπέρ και μία κατά. Εγκρίνεται επομένω. Και τώρα προχωρώ στο ψήφισμα. Παράγραφος 1, τροπολογία 5. Ναι, τροπολογία 5, σωστά. Γκέρ Μπράντι και Ντε Γιόγκ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Να βρω μια στιγμή την λίστα ψηφοφορία στη δική μου. Με συγχωρείτε μια στιγμή. Κάπου είναι εδώ. Κάπου εδώ είναι. Ίσως χρειαστεί κάποιο να μου δώσει. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ. Λυπούμε για την μικρή διακοπή. Τροπολογία λοιπόν 5, αυτή επαληθεύεται ηλεκτρονικά πέρα της ψήφου. ...15 ψήφοι υπέρ και 11 κατά, άρα εγκρίνεται. Ακολουθεί. Αφού εκπίπτει η 6, ακολουθεί η 4, δική μου, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7, Έπινγκ, Σαρνέκη κλπ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή. Παράγραφος 2. Τροπολογία 10. Σέντερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8 και 9. Ταυτόσημες. Μπορούν να ψηφιστούν μαζί. Α, όμως εκπίπτουν διότι εγκρίθηκε η 10. Ε, ο Κρι τώρα με την 11 υπέρ. Κατά επαλήθευση, επαλήθευση του κυρίου Ντέιβις υπαριθμών 11. Μου φαίνεται ότι απορρίφθηκε, πάντως τώρα τελείωσε η ψηφοφορία, 9 ε, ναι, υπέρ 17 κατά. 13 για Λασέντερ υπέρ, κατά. Απογές, εγκρίνεται. Η 12 εκπίπτει, 14 δική μου υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 15 έπιν και τα λοιπά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 16 δική μου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 Γκέρο Μπράντι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18. Ερενχάουζα υπέρ. Κατά. Αποχές. Μου φαίνεται ότι είναι τόσο κοντινό το αποτέλεσμα. Ας την επαληθεύσουμε. Τέλος. 13 υπέρ 14 κατά. 19 δική μου υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας την επαληθεύσουμε ωστόσο. Τέλος. 15 υπέρ, 12 κατά. 20. Γκρέσλε. Έχετε και προφορική. Α, άρα προφορική στο τετράγωνο. Αντί European Council and the Member States πρέπει να λέει European Council Member States. Λοιπόν, πρόκειται για προφορική τροπολογία, επί της προφορικής τροπολογίας. Η κυρία Γκρέσλη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 δική μου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 δική μου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται ουδής διαμαρτύρεται καλά τότε εγκρίθηκε λοιπόν 25 πάλι του κυρίου Έρενχάουζερ υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 26 υπέρ κατά. Μάλλον υπέρ ακόμη. Κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 20... Α, καλά, ας κάνουμε επαλήθευση λοιπόν για την 26. Πέρας. 16 υπέρ, 11 κατά. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 δική μου υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Α, με συγχωρείτε. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Είναι το 29. Αγιάλα Σέντερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30. De Jong και Sondergaard με προφορική τροπολογία της κυρίας Γκρέσλε, Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31, δική μου, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας προχωρήσουμε σε επαλήθευση. Τέλος, 12 υπέρ, 15 κατά. 33, Μάρτιν Έρενχάουζερ υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ο, 38 τώρα, κυρίας Αντρέασεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 δική μου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 Αντρέασεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 τώρα εισηγητής υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές. Πολύ, ε, πολύ κοντινό το αποτέλεσμα, δύσκολο να το διακρίνει κανείς, την επαληθεύουμε, παριθμό 41, πέρας, 15 ψήφοι υπέρ, 11 κατά εγκρίνεται. Το οποίο σημαίνει Πρέπει να ψηφίσουμε την 24 όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ, κατά, αποχές. Την παράγραφο δηλαδή 24 εγκρίνεται. 42 ε, τώρα δική μου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 δική μου υπέρ τροποποιήθηκε όμως προφορικά από την κυρία Γκρέσλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 ψήφι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται 46 της κυρίας Ματιού και της κυρίας Κρέσλε σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 48 δική μου υπέρ, κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Αλλά μιας και είναι δική μου, προτιμώ να είμαι απόλυτα ουδέτερος. Τέλος. 15 υπέρ, 11 κατά. 49 τώρα, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παριθμόν 50. Γκερμπράντι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτή. 51. Καλύπτεται από την 50, αλλά απορρίφθηκε η 50, οπότε ψηφίζουμε την 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται και αυτή. 53, Davis υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55, έπιν και λυπή υπέρ, κατά Αποχές. Ελάχιστη διαφορά. Ας το επαληθεύσουμε. Τέλος. Ψήφι 15 υπέρ 10 κατά εγκρίνεται. 56 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 Ερενχάουζερ υπέρ κατά αποχές Πάλι η διαφορά είναι πολύ μικρή. Ας επαληθεύσουμε. Πέρας. 14 υπέρ και 11 κατά. Άρα εκπίπτει 58. Ερχόμαστε στην 59 της κυρίας Τσέσκοβα υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται 60 Τσέσκοβα πάλι υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται και αυτή. Ακολουθεί η συμβαστική τροπολογία. Υπάρχει μόνο ένα ψήφι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 62-64 εκπίπτουν, 65 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 66, κυρίες Ματιού, Γιόν και Γκρέσλε, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 67 Ντε Γιόν κλπ. υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται αυτή 68 γκρέσλι υπέρ κατά αποχές ας αφήσει η διαφορά ας επαληθεύσουμε τέλος της ψηφοφορίας 15 υπέρ 11 κατά 69 γκρέσλε υπέρ κατά αποχές από την έδρα μου είναι δύσκολο να διακρίνω τη διαφορά ίσως όμως είναι η ίδια πλειοψηφία 15-11 μου φαίνεται θα είναι μου φαίνεται και όντως 15-11 70 δική μου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 μακοβέ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 Ανδρέας είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 Μακοβέ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 Ερενχάουζερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται αλλά ας υπαλληθεύσουμε 76 λοιπόν, Sondergaard de Jong. Πέρας. 20 προς 6. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79. Έπινς, Τσανέκη και λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 77. Σόντεργαρτ, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 78 δική μου, υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 82 δική μου, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 έπινκ και λοιπόν υπέρ κατά άποχες ασαφές το αποτέλεσμα νομίζω αν είναι δυνατόν να σηκώνει τα χέρια πιο ζωηρά επαληθεύουμε λοιπόν Πέρας. 23 υπέρ, 4 κατά. 84 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85 Τσέσκοβα υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 Τσέσκοβα υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89 Έπινγκ και λοιπόν υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 88 βαντάλιν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 Αντρέασεν με προφορική τροπολογία της κυρίας Γκρέσλε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 Βαντάλεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 Μακοβέ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92 Μακοβέ πάλι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. 93 Τεγιόν και λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94 Τελάνγκια υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 Βαντάλεν υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 96 έπιν και υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 δική μου υπέρ Α, Ας επαληθεύσουμε την ψηφοφορία της 98. Τέλος. Απερίφθη με μεγάλη διαφορά. 3 υπέρ, 23 κατά. Για και μπράβο. 99 δική μου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100. Κρέσλε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 101. Ανδρέασεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 Ανδρέας είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 Τσέσκοβα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 δική μου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 Βαντάλεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 Γκερμπράντι και λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 Ματιού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 108 Ερενχάουζερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτή τελική ψηφοφορία παρακαλώ ονομαστική Τέλος. 24 υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν κυρία Συγητρία. Κύριε Σκερπράντη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγκρίναμε την τροπολογία 5 και προσπαθούμε τώρα, ε, ζητούμε μια ξεχωριστή συζήτηση τον Απρίλιο στην Ολομέλεια για την απαλλαγή του Κοινοβουλίου. Και πέρυσι το κάναμε αυτό με ένα ψήφισμα στο Κοινοβούλιο. Ξέρω όμως ότι η διάσκεψη των Προέδρων τον περασμένο μήνα αποφάσισε να μην γίνει κάτι τέτοιο για να αποφύγουμε να βρεθούμε στην περίεργη κατάσταση η Ολομέλεια τον Απρίλιο να κάνει συζήτηση. Δηλαδή, θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο της Επιτροπής να αποστείλει μια επιστολή στη διάσκεψη των Προέδρων, αν γίνεται, να επαναλάβουμε αυτό το αίτημα, να το τονίσουμε και να ε, επισυνάψουμε και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εδώ στην Επιτροπή μας. Μάλιστα. Ε, κατάλαβα τι ζητήσατε, κύριος Γκάιερ. Νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε τέτοια πράγματα. Θα θυμάστε στην τότε ημερήσια διάταξη για την Ολομέλεια Είχαμε ε, προβλέψει χωριστή ε, συζήτηση. Εγώ έχω άλλη πληροφόρηση από σένα. Και η συγγήτρια κυρία Ορτής ε, ζήτησε χωριστή ψηφοφορία για το Κοινοβούλιο και μάλιστα ειδική συζήτηση για αυτό το θέμα. Άρα το επιβεβαιώνει η συγγήτρη αυτό. Ε, η γραμματέας μου λέει ότι ε, αυτά που ισχυρίζεται ο κύριος Γκάιερ ισχύουν. Σας ικανοποιεί αυτό κύριε Γκεμπράντη. Μα αυτό είναι ακριβώς το θέμα. Κάθε χρόνο αυτό κάνουμε. Είναι μια γενική συζήτηση, αλλά η τροπολογία 5 ζητεί ξεχωριστή συζήτηση ε, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή αν προεδρεύει ο κύριος Μάλτιν Σούλτς έτσι ώστε και δημόσια να διατρανωθεί αυτό. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γι' αυτό κάναμε και την τροπολογία, να ε, αναλάβει τις ευθύνες για τον προεπολογισμό ε, του Κοινοβουλίου. Όχι κοινή συζήτηση, ξεχωριστή, έκτακτη, ειδική συζήτηση για το Κοινοβούλιο. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα. Και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες δεν έχει εγγραφεί έτσι στην ημερήσια διάταξη. Μάλιστα, καλώς. Η κυρία Γιάλα Σέντερ θέλει το λόγο. Ναι, το μόνο που θα ήθελα είναι να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα για να μην είναι αντιφατικό και για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα να ζητήσουμε τα ίδια. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην μας στείλουν τον κύριο σε μετά, αλλά να έρθει ο κύριος Μπαρόσο, πρόεδρος, υπόλογος. Και ε, για το Συμβούλιο ακριβώς τα ίδια. Να μην μας στείλουν κάποιον άλλο, να έρθει αυτοπροσώπως η Προεδρία. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι. Να μην είμαστε εμεί βασιλικότεροι του βασιλείου, μάλλον παπικότεροι του Πάπα, τώρα που έχουμε και νέο Πάπα. Εκτό από τον κύριο... Ναι κύριε Γεβράντη, σα έχω δει. Ε, θα σα δώσω το λόγο γιατί εσεί το εμπνευστή της όλης ιστορία. Ναι. Μου δίνει το προσωπικό τώρα την τελευταία ημερήσια διάταξη που έχει πάλι αλλάξει ε, σε σχέση με την προηγούμενη το σχέδιο και τώρα πραγματικά προβλέπεται ξεχωριστή συζήτηση. Έχει δίκιο ο Γιάννης Γκάιερ. Όντως, έχει εγγραφεί στη ημερήσια διάταξη. Ζητώ συγγνώμη για την παρεξήγηση. Αντίθετα, εγώ πιστεύω ότι εάν πρέπει να συζητήσει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, δεν πρέπει να προεδρεύσει. Maar dan heb je ondervoorzitters. Έχουμε και την Προέδρου, ξέρετε, για αυτή τη δουλειά. Eh, eh, Ο κύριος Γκερμπράντι έκανε μια ερώτηση. Ε, νομίζω ότι τώρα ικανοποιήθηκε με την απάντηση που του δόθηκε και θεωρούμε λήξαν το θέμα. Εντάξει, μπορούμε να περάσουμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Τελευταία για σήμερα παρακαλώ. Έτσι δεν είναι, πολύ ωραία. Το σημείο 7. Είναι η έκθεση του κυρίου Κάλφιν. Θέλετε το λόγο παρακαλώ. Δεν τον βλέπω. Α, να, εδώ είναι ο κύριος Κάλφιν. Ναι, παρακαλώ. Θέλετε το λόγο. Πάρα πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Στην Επιτροπή μου ψηφίσαμε ε, για την Επιτροπή Εξωτερικών ε, Εξωτερικής Δράσης, καθώς επίσης και για κάποιες άλλες ε, διαδικασίες. Εδώ δεν είναι η ψηφοφορία για την απαλλαγή, αλλά για την αντιμετώπιση από την ΑΠΦΕΤ, που είναι η αρμόδια καθήλια Επιτροπή του θέματος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Εδώ θα έχουμε και τα δύο έγγραφα, δηλαδή και την απαλλαγή, καθώς επίσης και την, ε, την έκθεση, καθώς επίσης και την θέση της Επιτροπής μας εδώ, του τι θα γίνει στο μέλλον. Επίσης αναφέρεται και στην, στον κατάλογο της ψηφοφορίας, αλλά... Οι τροπολογίες 1, 3, 4 και 5 την χάνουν τη στήριξή μου. Οι τροπολογίες ε, Γκρέσλε νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να έχουμε κάποιες ελαφρές τροποποιήσεις στο κείμενο βάσει προφορικών τροπολογιών. Ευχαριστώ. Okay. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κάλφιν. Ναι, και εγώ, εγώ είχα μπερδευτεί. Δεν είναι η ίδια η απαλλαγή, είναι μια σύσταση. Ε, παρατηρήσεις έχουμε? Όχι. Ωραία, ας ψηφίσουμε τότε. Τροπολογία παριθμών 1. Της κυρίας Γκρέσλε. Υπέρ. Δικιά σας τροπολογία. Νομίζω μπορείτε και να την υπερψηφίσετε ακόμα, κυρία Γκρέσλε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 2, Γκρέσλε υπέρ. Κατά. Άποχες. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Ας το ελέγξουμε όμως. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 και πάλι της κυρίας Γκρέσλε. Υπέρ. Κατά. Α, ναι, με την προφορική, εντάξει. Ε, ε λοιπόν, τροπολογία 3 με την προφορική της κυρίας Γκρέσλε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 4 της κυρίας Γκρέσλε με προφορική του εισηγητού υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 5 με την προφορική πάλι του εισηγητού επί της τροπολογίας Γκρέσλε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και εδώ τελειώσαμε τις τροπολογίες ηλεκτρονικά θα κάνουμε την τελική ψηφοφορία Εσ... Ομόφωνα εγκρίνεται κύριε Κάρφιν και συγχαρητήρια. λοιπόν ολοκληρώνονται οι σημερινές εργασίες. Και έχετε μία ωρίτσα για πάτε να πιείτε κάτι. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 9. Wow, what efficiency.